πρακτικά τις 26ης ε, και 27ης ε, συνόδου έχουν δημοσιευτεί, δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσεις. Για τα πρακτικά. Περιμένετε, περιμένετε. Για τα πρακτικά θέλετε να πάρετε το λόγο. Εκτός μικροφώνου μιλητής. Ah, για τα πρακτικά θέλετε το λόγο. Όχι. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Καταρχά, θα πρέπει να πω κατά πόσο υπάρχουν αντιρρήσει για τα πρακτικά. Δεν ξέρω, υπάρχουν πρακτικά για τα, ε, αντιρρήσει για τα πρακτικά. Όχι. Ε, ωραία, λοιπόν. Εκεί κυρώνονται θέλετε ένα διαδικαστικό ζήτημα να θέσετε. Έχετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε, στο όνομα όλων των βουλευτών του Πέντε Αστέρων θέλω να τονίσω το σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται ο κύριος Ρενάτο Σόρμπο και από τους σοσιαλιστές και άρα ολόκληρο το Ευρωκοινοβούλιο. Τρία 6.2 του κανονισμού κώδικα διοντολογία και συμπεριφορά των βουλευτών. Γιατί αυτός ο κύριος καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση για φοροδιαφυγή και ωστόσο εξακολουθεί να είναι πλήρω μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων που ακριβώ αποφασίζουμε για θέματα φοροδιαφυγής και φοροαπάτης. Βρισκόμαστε ενώπιον μια γιγάντιας σύγκρουσης συμφερόντων με την εντολή μα, με τη θητεία μας μάλλον, που μας δεσμεύει για διαφάνεια. Και σα ζητώ Πρόεδρε να τα επαληθεύσετε αυτά που σας είπα και να προβείτε στα απαραίτητα διαβήματα και ζητώ αμέσως από τον κύριο Σόρμπο να παραιτηθεί αμέσως, από τον κύριο Πιτέλα να επιβλέψει την ομάδα του, να ελέγξει τι συμβαίνει, γιατί εδώ δεν μπορεί να εξακολουθεί αυτή η κατάσταση εντός του Ευρωκοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ να διαφυλάξετε την αξιοπρέπεια αυτή τη αίθουσα και αυτού του θεσμού. Δεν μπορεί να κάθεται εδώ στα ίδια έδρανα ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή. Ηρεμήσατε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Μάλιστα. Όχι κύριε Πιτέλα. Δεν θα ξεκινήσουμε συζήτηση για το θέμα αυτό. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει κράτος δικαίου, ξέρετε δεν ήταν αντιδικαστικό αυτό, ήταν πολιτική δήλωση. Ο συνάδελφος που αναφέρεται καταδικάστηκε ε, και υπέβαλε έφαση κατά της δικαστικής απόφασης και μέχρι να υπάρξει η δευτεροβάθμη απόφαση ε, σεβόμαστε το κράτος δικαίου και δεν έχω ως πρόεδρος καμία διάθεση και καμία εξουσία να επέμβω. Αυτό εναπόκειται στην Ιταλική δικαιοσύνη. Υπάρχει η ασυλία των βουλευτών, άρτικη ασυλία του βουλευτή. Δεν είχαμε να κάνουμε κάτι άλλο και θα ακολουθήσει λοιπόν το δρόμο της Ιταλική δικαιοσύνη. Καταλαβαίνω και κατανοώ ότι ως πολιτικός θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα πρακτικά για να κάνετε αυτή την μονομερή δήλωση. Ο κ. Φιλιπ και ορίστηκε από την Μελγική Κυβέρνηση και ο κ. Γιάννος και οι δύο λοιπόν αυτοί οι βουλευτές ορίστηκαν, διορίστηκαν στο ρεκτικό συνέδριο. Και τους συγχαίρω και πλέον λοιπόν η θέση τους είναι καινέ ε, με τις αποφάσεις